Dear colleagues, uh, welcome once again. Και πάλι καλώς ήρθατε συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος. Ας αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Να είστε σίγουροι ότι θα βάλετε στη σχισμή την κάρτα σας και ξεκινούμε με το 12, 13, 14 και 28. Θα γίνει με ενιαίο τρόπο η ψηφοφορία. Κυρία Βίκστρομ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε να πω δύο λόγια πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Γιατί όπω γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε ο τρίμηνο διάλογο για αυτό το θέμα την άνοιξε Και τώρα, μετά από σκληρή δουλειά των συνεργατών μα εδώ στο Κοινοβούλιο, ολοκληρώσαμε μια μορφή του κειμένου την οποία θα ψηφίσουμε. Αυτό που έχουμε τώρα δεν είναι για το σήμα κάποια επανάσταση, είναι ένα εξηγανισμό αντίθετα το οποίο ήταν και ο στόχος μας. Ήδη υπάρχει ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί εύρεμα και απλώς χρειαζόταν ε, κάποιες πινελιές, χρειαζόταν να λαδοθεί λίγο το σύστημα για να είναι ακόμα πιο εύρεθμο για τώρα και για το μέλλον και με αυτή την αλλαγή τώρα θα αναβαθμίσουμε το θέμα των σημάτων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, επίπεδο, ε, λιγότερο κόστος, καλύτερο για τους χρήστες, και ε, πιο πολύ θωρακισμένο, ε, θα κατοχυρωθεί και η ελευθερία της έκφραση. οπότε επίση τώρα θα έχουμε καλύτερη δομή στη διακυβέρνηση όσον αφορά την, την υπηρεσία για τα σήματα και τώρα θα ονομάζεται το Γραφείο πνευματική ε, Ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πιο σωστό όνομα και τώρα είπαμε ότι το κεντρικό μας ενδιαφέρον είναι οι χρήστε Καταφέραμε λοιπόν να τους καλύψουμε και επίσης θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους και του ηγητές όλο μας το επιτελείο, όλους τους παλιούς του Κοινοβουλίου, όλους που ήρθαν για αυτό το δύσκολο θέμα και επίσης να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ακάματα μας βοήθησε και προσπάθησε να γεφυρωθούν οι διαφορές των δύο θεσμικών οργάνων για αυτό το περίπλοκο πακέτο διατάξεων και επίσης ευχαριστώ και όλους από όλες τις Προεδρίες του Συμβουλίου με τους οποίους συνεργάστηκα. Ήταν φανταστικό να συνεργαστούμε με την Λουξεμβουριανή Προεδρία για όλα αυτά τα ζητήματα και ολοκληρώθηκε η υπόθεση την Άνοιξη. Και πρέπει να ευχαριστήσω και την Ιταλική και την ε, Λετωνική Προεδρία για τις προσπάθειές τους ε, στην τελική ευθεία. Αλλά βέβαια θα πρέπει και τους συνεργάτες μου να τους ε, ευχαριστήσω ιδιαίτερως γιατί δουλούσαν σκληρά. Ήταν ε, μια μακρά διαδρομή, πολλά χρόνια και τώρα φτάσαμε στον τερματισμό. Ας ψηφίσουμε. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε το σημείο 12 ηλεκτρονικά. δεν uh, Open the vote We are missing one person. Κάποιος λείπει. Okay. Uh, uh Και εγκρίθηκε 21. 2. Πάμε τώρα στο 13. Electronically, Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για το δεύτερο σημείο. I close the vote. Πέρας ψηφοφορίας. Adopted. Εγκρίνεται. 14. Ψηφίζουμε. I close the vote. περα ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Συμπαθάτε με λέει ο πρόεδρος. Ξέχασα να δώσω για αυτό το θέμα τον λόγο στον κύριο Σάιερ. Τώρα για το 28 κύριε Σβιέφκα θέλετε το λόγο. Κυρία Χάουταλα. Απλή κωδικοποίηση. Κανένα πρόβλημα. Δεν είχαμε μετάφραση στα κροατικά, αυτό ήταν ένα πρόβλημα να ψηφίσουμε σήμερα. Προτείνω γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει Σέγγεν την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, ωραία, λέει ο πρόεδρο. Ψηφίζουμε. Close the vote. Πέρασε Εγκρίνεται. Κύριε Χρυσόγωνε, συγγνώμη γιατί ξέχασα να σας δώσω το λόγο. Κύριε Άντερσον, να σας πω ότι παρίσταμε, αλλά δεν έχω την κάρτα μου. Λέει ο κύριος Άντερσον. Θέλει να καταχωρήσουμε τη θετική ελληνική ψήφο. Άντερσον. Θα ψήφισε το ίδιο όπως και η Χάιντι. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ακριβώς σε ποιο σημείο είμαστε. Η κυρία Χαούτα, λεκτό μικροφώνου λέει ψήφισε ναι αλλά δεν μπορώ να το κάνω εγώ για σένα. Συνεχίζουμε την ψηφορία λέει ο Πρόεδρος. Για την έκθεση που αφορά την πράξη ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο κ. Τζαμπάσκι θέλει το λόγο πριν ψηφίσουμε. Όχι. Όχι, θα ψηφίσουμε. Ωραία, θα ψηφίσουμε δυνατά στις χειρός λοιπόν. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά καλύτερα να το τσεκάρουμε να το ελέγξουμε λοιπόν Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 90. Απορρίπτεται. Τροπολογία 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 2 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν γιατί δεν είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Απερίφθη. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Τροπολογία 58, 78 ε, υπέρ. Συγγνώμη, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Δεν υπάρχει δεύτερο τμήμα, λέει ο πρόεδρος τελικά. Δεύτερο τμήμα υπάρχει τελικά, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 60, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 65, υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 69 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 σε 3 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117. Και εδώ υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε το σημείο με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Θέλω να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 150 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απερίφθη. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 149. Ναι, απερίφθη. Συνεχίζουμε. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 151. Συμβιβασμός 11 μάλλον λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 183. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τροπολογία 186. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 178. Χωρίς την προφορική τροπολογία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Και τώρα ψηφίζουμε με την ε, προφορική τροπολογία το ίδιο κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 70 με την προφορική τροπολογία. Με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα, χωρίς την προφορική τροπολογία, την 170 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά ε, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ να κάνουμε για αυτό το σημείο. Εγκρίνεται. Ενώ εγώ είχα την αίσθηση ότι είχε απορριφθεί. 188 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα θα ψηφίσουμε διονομαστικής κλίσεως επί του συνόλου άρχεται Yes, τη ψηφοφορία. ψηφοφορίας ενεκρίθη. Συγχαρητήρια κύριε Τζαμπάσκη. We continue. Συνεχίζουμε με το σημείο 16. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών. Ανακοινώνουμε λοιπόν ότι ο κύριος Χρυσόγονος ορίστηκε εισηγητής για μια ε, έκθεση εφαρμογής της ε, Ευρωπαϊκής Εντολής Πληρωμής. Ο κύριος ε, Μάστερκαν είναι εισηγητής για μια γνωμοδότηση τη συμφωνία σχετικά με τη συνεργασία ανάμεσα στη Eurojust και στην Ουκρανία. Ορίζονται οι εξής μόνιμοι εισηγητές για τους έξι μήνες από την πρώτη πρώτου δέκα 16. Κύριος Φως για την νομική βάση. Ο κύριος Λεμπρετό για την επικουρικότητα. Ο κύριος Τζαμπάσκι για τα ε, ζητήματα κομματολογία και πράξεις κατά εξουσιοδότηση και η κυρία Φεράρα για την κωδικοποίηση και τις αναδιατυπώσεις. Συνεχίζουμε με το σημείο 17, έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετήσια έκθεση για το 2014. Το λόγο έχει η κυρία Χάουταλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μια ετήσια έκθεση και προσπαθούμε να συντονίσουμε τα πράγματα και να ορίσουμε το χρονοδιάγραμμα παράλληλα με την ετήσια έκθεση σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Είναι διαφορετικά πράγματα βέβαια, όμως τα εξετάζουμε μαζί έτσι ώστε να μας δώσουν μια γενικότερη εικόνα. Ε, σας παρακαλώ, λέει ο να κάνετε ησυχία, ιδιαίτερα όσοι μιλάτε στους διαδρόμους. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα λοιπόν από την αρχή. Προσπαθούμε να συγχρονίσουμε την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με εκείνη για την ε, εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Ο κύριος Κάριμ έχει αναλάβει αυτές τις εκθέσεις. Συνήθως με αυτές τις εκθέσεις το Κοινοβούλιο ασκεί έλεγχο στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση τα καθήκοντά της ως θεματοφύλακα των συνθήκων. Ακόμα και αν η σωστή εφαρμογή ε, της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν πρέπει να παραμένουμε σε αυτό, αλλά και να ελέγχουμε το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της. Ένα σχόλιο που μπορούμε αρχικά να κάνουμε είναι κάτι που δεν είναι καινούριο και είναι πραγματικά περίεργο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αντιδράσει μέχρι τώρα. Οι επίσημες διαδικασίες επί παραβάση μειώνονται. Ο αριθμός των πιλωτικών, όπως λέγονται, ε, θεμάτων αυξάνεται αντίθετα. Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς ε, ασκεί τα καθήκοντά της λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ω θεματοφύλακα των συνθήκων και δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτήν την περίπτωση είναι αρκετά ε, διάφανη ή ε, λειτουργεί υπέρ των συμφέρων ε, των ενδιαφερόμενων μερών. Η Επιτροπή αυτή λοιπόν ζητεί την πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την πιλωτική διαδικασία της Ένωσης και τις εκκρεμής υποθέσεις. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή mm-hmm. αρχίσει μια διαδικασία επί παραβάση και προτού ε, αρχίσει να εργάζεται σε πιλωτικά ε, θέμα, προγράμματα. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να έχουμε πρόσβαση στο πιλωτικό πρόγραμμα και υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι ότι υπάρχουν τρεις συνδεδεμένες χώρες, η Ουκρανία, η Μολδαβία και η ε, Γεωργία. Και όπως γνωρίζετε καλά, κύριε Πρόεδρε, όταν πήγαμε με την Επιτροπή Ίντα στην Ουκρανία, είδαμε ότι αυτές οι χώρες βρίσκονται στη θέση να πρέπει να μεταφέρουν περίπου 300 έως 400 νομοθετικές ε, πράξεις μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να αρχίσουμε να ελέγχουμε το πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές θεσμικές αδυναμίες σε αυτή τη χώρα, σε αυτές μάλλον τις χώρες, ας πούμε λόγω της ε, πολιτικής εκατάστασης των πολιτικών ε, σωμάτων του εκλεγμένου κοινοβουλίου και γνωρίζουμε επίσης πως υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στο δικαστικό σύστημα των χωρών αυτών. Οι χώρες βέβαια αυτές έχουν δεσμευτεί να κάνουν μεταρρυθμίσεις μέσω, ε, στα πλαίσια της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Για πρώτη φορά προσπαθούμε να διερευνήσουμε το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσει η εφαρμογή και η μεταφορά αυτών των νομικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα γίνει σωστά. Και να αναφέρω επίσης ότι τα κοινοβούλια των ε, τριών αυτών ε, χωρών εκτίμησαν το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε αυτήν την θέση να δημιουργήσει νέες συνεργασίες με αυτά έτσι ώστε να τα βοηθήσει στην μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας διότι όπως ε, ξέρουμε όλοι ο νομοθέτης πρέπει να εγκρίνει και να περάσει αυτούς τους νόμους. Τρίτον, να αναφέρω ότι μέρος του προβλήματος της έλλειψης διαφάνεια της διαδικασίας επί παραβάση και της επιλοτικής διαδικασίας οφείλεται στην, στον έλεγχο της ε, διοικητικής διαδικασίας όπως αναφέρετε και εσείς κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο έκθεσης που θα εξετάσουμε αμέσως μετά στην ημερήσια διάταξη είναι πολύ σημαντικό. Επίσης είναι σημαντικό οι ελλείψεις που παρατηρούνται στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και σχετίζονται με τις επιδόσεις της Κομισιόν αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων οφείλονται σε αυτές τις παρατυπίες στη διοικητική διαδικασία. Η ομάδα εργασίας που συστάθηκε με επικεφαλή σε αυτήν την Επιτροπή βρίσκεται στη θέση στις 11 Ιανουαρίου να παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης και να διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου ένας ευρύτερος διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένη για την, από την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει και από την γραμματεία και από τον ε, ερευνητικό κλάδο. Πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτός ο κανονισμός θα φέρει πράγματι προστιθέμενη αξία στις επιδόσεις της και να πω επίσης ότι ίσως θα μπορούσε να αντικαταστήσει πολλές σελίδες της ε, καλύτερης νομοθεσίας. Ήταν ένα ε, συλλογικό έργο ανέκαθεν, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι ελπίζω στην συμμετοχή όλων από εσάς και πέρυσι όταν ήταν εισηγητής ο κύριος Χρυσόγονος προσέθεσε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούσαν το πρόβλημα της ελιτότητας και τη σχέση του με την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορούμε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό, να δούμε λίγο ε, πιο κοντά την κατάσταση. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η χάρτα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που βρίσκεται αγκυροβολημένη στις συνθήκες είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά. Γι' αυτό λοιπόν ίσως μπορούμε να διερευνήσουμε και αυτήν την πτυχή της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελβό έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να μιλήσω και λογαριασμό της κυρίας Κάφνου που δεν μπορέσε να παραστεί και μου έχει δώσει εδώ αυτά τα οποία είχαν παρατηρήσει, θα σα διαβάσω ή στα γερμανικά. Κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, η Σίλβια Κάουφμαν θα ήθελε να αναφερθεί σε δύο σημεία τα οποία θεωρεί σημαντικά για την έκθεση. Καταρχά, ε, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ο αυξανόμενο αριθμό τη ε, μη εφαρμοσμένη ε, νομοθεσία τη Ένωση από τα κράτη-μέλη. Το 2014 υπήρξαν 1.347 εκκρεμίσεις διαδικασίες επί παραβάσεις. Και πολλές φορές τα κράτη-μέλη ε, καθυστέρησαν στην έναρξη νέων ε, νέας, ε, στην εφαρμογή νέας νομοθεσίας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, όμως το πώς θα το κάνουμε παραμένει προβληματικό. Τα κράτη-μέλη όταν δεν πληρούν τις ε, υποχρεώσεις τους οδηγούν σε αυτά τα προβλήματα και δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση. Η μη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής ενομοθεσίας οδηγεί de facto σε διάκριση εις βάρος των πολιτών και σε αστάθεια στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη-μέλη είναι ε, υπεύθυνα για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ανομοθεσίας και τη μεταφορά του στο εθνικό δίκαιο και πρέπει να πληρούν αυτές ε, τις προϋποθέσεις και να τηρούν τις υποσχέσεις τους και τις υποχρεώσεις τους. Στο χέρι μας είναι να δούμε πόσο μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία εφαρμογής και μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Οι διαπραγματεύσεις ε, ανάμεσα στα θεσμικά όργανα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως ε, και τόνισε άλλωστε ναι. και ο κύριος Φερχόφσταν στην τελευταία συνεδρίαση. Είναι ε, αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα νέο όργανο εφαρμογής της νομοθεσίας. Έπειτα, το δεύτερο πρόβλημα είναι το λεγόμενο gold plating, που χρειάζεται, από ό,τι φαίνεται, ένας σαφής ορισμός για το τι σημαίνει αυτό. Η δική μας ομάδα έχει ε, την άποψη ότι καταρχάς είναι αναγκαίο ότι σε όλα τα επίπεδα, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό και τοπικό, να αναλογιστούμε πόσο ε, μπορεί να μειωθεί ο ε, Διοικητικό ε, φόρτος και η γραφειοκρατία. Αυτό δεν πρέπει φυσικά να αμφισβητήσει το δικαίωμα που έχουν τα κράτη-μέλη ε, να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να δημιουργήσουν ενδεχομένω υψηλότερα πρότυπα που θα αποτελέσουν καλό παράδειγμα για τη συνέχεια. Σίγουρα πρέπει να μειωθεί το διοικητικό άχθο και αυτό θα γίνει μόνο με πολιτική βούληση. Είναι κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη και πρέπει να αφήσουμε στο κάθε θεσμικό όργανο να έχει τις δικέ του αρμοδιότητε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Βιέσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Και κάθε χρόνο οδηγούμαστε στα ίδια συμπεράσματα. Πολύ λίγα γίνονται όμως αφού γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση της ε, κυρία Χάουταλα, που είναι πάρα πολύ καλή, με πολύ ε, σωστές προτάσεις, ιδιαίτερα σχετικά με το διοικητικό δίκαιο και ε, το, τις εργασίες μας, το πώς θα εργαστούμε, <clears throat> πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Και ελπίζω να επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες είναι αναγκαίες πιστεύω. Το βλέπουμε κάθε μέρα εξάλλου. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Κάθε χρόνο βέβαια το λέμε, έχουμε ένα μέσο συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό το μέσο μας συνδέει. Μπορούμε να συζητήσουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια για τους λόγους που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα προβλήματα έγκαιρης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στα εθνικά συστήματα, στην εθνική νομοθεσία. Ίσως η συνεργασία λοιπόν μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ο σωστός τρόπος για να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση. Δεν θα βελτιωθεί βέβαια σημαντικά, το γνωρίζουμε αυτό, όμως πρέπει να πω ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη προσεγγίζουν το ζήτημα αυτό κατά το δικό τους συμφέρον και κατά πόσο τους συμφέρει η σχετική νομοθεσία. Εάν ένας ευρωπαϊκός νόμος συμφωνεί με, τις, ε, με τα εθνικά συμφέροντα θα τον μεταφέρουμε. Διαφορετικά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καθυστερήσουμε τη διαδικασία ή για να μην μεταφέρουμε καθόλου την νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο. και προσπαθούν τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν ε, τις αδυναμίες ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στους πολίτες της. Αυτό έγινε στην περίπτωση των ε, κεριών και, του, και της εφλόγας από τα κεριά. Ένα παράδειγμα μόνο σας δίνω. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε έντονα από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν σαφή και η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και περιέχει πολύ σημαντικά στοιχεία. Ωστόσο, πιστεύω ότι το επόμενο έτος όταν θα συζητήσουμε την εφαρμογή της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το 2015 η συζήτησή μας θα είναι πάνω κάτω η ίδια. Όμως ελπίζω να μπορέσουμε να αναφέρουμε πως έχει υπάρξει κάποια βελτίωση. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητά το λόγο, λέει ο πρόεδρο. Ήθελα να προσθέσει κάτι κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τους, ε, για τα σχόλιά σας. Και θα συζητήσω με την κυρία Κάουφμαν για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συζήτηση αυτή για τα νέα μέσα που πρότεινε που θα βελτιώσουν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι κάπως ε, να φανταστώ ποια θα είναι αυτά, όμως πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα τις δυνατότητες που έχουμε. Σίγουρα βέβαια πρέπει και να λάβουμε υπόψη αυτήν την επιχρήσωση, το gold plating που λέμε. Αναφέρθηκε Επίσης ε, στην έκθεσή της ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες που δεν έχουν εξεταστεί από το Κοινοβούλιο. Ειδικά το θέμα του gold plating αναβάλλεται και δεν γνωρίζω γιατί. Κύριε Διεύκα, μας μιλήσατε για την πολιτική διάσταση του θέματος και το συμφέρον που έχουν τα κράτη-μέλη μας αναφέρεται και αυτό το παράδειγμα με τη φλόγα από τα κεριά. Θα δούμε λοιπόν ε, τι συνεργασία θα μπορούσαμε να έχουμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να αναφέρω μόνο ένα θέμα που σχετίζεται με τις ε, τρεις ε, χώρες που αναφέρατε, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία. Σίγουρα υπάρχουν, ε, υπάρχει Κόσακ, που είναι ένα φόρουμ αρκετά ε, διακοσμητικό ίσως θα έλεγα και το λέω επειδή ήμουν μέλος της ΚΟΣΑΚ. Δεν είναι τόσο πρακτικό μέσο για την ε, εφαρμογή της ε, επικοινωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη συνεισφορά όλων σας από όλες τις ομάδες με το σκεπτικό να δημιουργήσω ένα σχέδιο έκθεσης Ιανουάριο ή Φεβρουάριο περίπου μάλλον τον Ιανουάριο, και να συζητηθεί στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο για να πάει τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Είναι μια σημαντική ευκαιρία, πιστεύω, αυτή, για να μην διαονίζεται αυτή η κατάσταση που ανέφερε ο κύριος ε, Σβιεύκα και για να μην καταλήξουμε του χρόνου να συζητάμε και να λέμε τα ίδια πράγματα. Πρέπει να βρούμε νέες λύσεις, λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χαρόταλα, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε με το σημείο 21. Συζήτηση για σχέδιο έκθεσης όσον αφορά την δημόσια πρόσβαση ή στα έγγραφα. Έχετε για άλλη μια φορά το λόγο κυρία Χαουτάλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω συντάξει ένα έγγραφο με πέντε σημεία. Όπως είπαμε και στην πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων για το ίδιο θέμα. Και τώρα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο ότι δεν έχει γίνει εφαρμογή του κανονισμού 1049 του 2001 όσον αφορά την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να καταγράφουν το, τα, τα έγγραφα και αν υπάρχει κάποιο μητρό. Πάρα πολύ σοβαρό κενό και έχουμε συνοηθεί σχετικά και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα πρέπει να υπάρξει αυτό το μητρό, αλλιώς δεν γίνεται οι πολίτες ή οποιοδήποτε άλλος να γνωρίζει σε ποια έγγραφα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να κάνει σχετική αίτηση και έχει πει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σημείο προσβασιμότητας, θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες και κριτήρια για το τι γίνεται με τα, με τα έγγραφα για να υπάρχει τελικά αυτό το μητρό, αυτό το πρωτόκολλο. Έχουμε μία διοργανική επιτροπή που είχε συγκροτηθεί από αυτόν τον οργανισμό τον 1049 σε σχέση με τα έγγραφα, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν ε, είναι και τόσο δυναμική. Γι' αυτό ακριβώς και για άλλους λόγους δεν έχει τηρηθεί σχετική δέσμευση όπως αυτή περιγράφεται από τον κανονισμό. Άρα θα πρέπει αυτή η Επιτροπή ε, να δουλέψει πιο εντατικά και να αναφέρει σχετικά όπου πρέπει. Τώρα κάτι άλλο το οποίο ε, αφορά διάφορα άλλα θεματολόγια είναι η νομοθετική διαδικασία. Γιατί υπάρχει μια περιομένη πρακτική για διοργανική συμφωνία όσον αφορά τους τρίμερες διαλόγους και τα νομοθετικά κείμενα και έχουν υπάρξει σχόλια από πλευράς του Ευρωπαίου Δησομεσολαβητή για το ότι το κοινό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα έγγραφα του τριμερούς διαλόγου. Όχι για να αμφισβητηθούν οι τριμερείς διάλογοι που είναι τόσο αποτελεσματικό μέσο εξέβρεσης λύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και άλλοτε βοηθά, άλλοτε βοηθά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά άπαξ και οι συνθήκες υποχρεώνουν τα θεσμικά όργανα να εξασφαλίσουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα για να μην μπούμε ένα σκοτεινό σημείο γιατί και γίνονται και κλεισμένων ε, αυτοί οι διάλογοι και δεν μπορεί κανείς να δει τα σχετικά έγγραφα. Βέβαια πολλές φορές κάποιοι προνομιούχοι αποκτούν πρόσβαση στα έγγραφα οπότε και βέβαια έχουν το πάνω χέρι και πλεονέκτημα των υπολείπων. Οπότε και εγώ παραλαμβάνω και την έκκληση του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει πριν από τη συμφωνία οι τριμμένες διάλογοι ε, να διέπονται από αυτή την αρχή της φιλελεύθερης πρόσβασης στα έγγραφα. Άρα να υπάρχει αυτή η διαφάνεια στην ουδετική διαδικασία γιατί έτσι αναβαθμίζουμε τη δημοκρατικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται ε, για το θεμέλιο κάθε νομοθετικής πράξης και άλλωστε έχουμε και απόφαση του Συμβουλίου. Έχουμε την υπόθεση της ε, Σουηδίας κατά ε, του Συμβουλίου Σουηδία και άλλη κατά του Συμβουλίου αφορούσε κάποια νομική γνωμοδότηση Ο δε διαμεσολαβητής έχει πει ότι Μπορεί να κάνει έρευνα η επιστροφή ε, για το τι γίνεται στους τριμμένους διαλόγους και κανένας ε, δεν ε, έχει αμφισβητήσει το δικαίωμα του διαμεσολαβητή στα, στα έγγραφα παρά κάποια προβλήματα που έχουν υπάρξει. Μπορεί όμως να εμπλακεί ο διαμεσολαβητής ή η διαμεσολαβήτρια σε αυτή τη διαδικασία που γίνεται μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Δεν λέω αυτό τώρα να το κάνουμε σημαία και να δώσουμε άγριες μάχες με τα άλλα θεσμικά όργανα. Γιατί είναι κατοχυρωμένο το δικαίωμα της πρόσβασης στα έγγραφα. Αυτό λέω και εγώ στην έκθεσή μου. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το Κοινοβούλιο να μην ε, υποστηρίξει το αίτημα της διαμεσολαβήτριας να στείλει κάποιον ε, υπαλληλό τη, ε, όπου τυχόν ενδιαφέρεται, να παρακολουθήσει τους τριμερείς διαλόγους, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα βέβαια της γνωμοδότησης, ε, το λέω γιατί είναι σχετικό. Υπάρχει το δικαίωμα της διαμεσολαβήτριας για πρόσβαση ή στα έγγραφα. Και έχω λόγους να πιστεύω ότι τελικά θα υπάρξουν από τη διαμεσολαβήτρια κάποιες συστάσεις όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους και τα έγγραφα καλά δεν μπορώ τώρα να μαντέψω πού θα καταλήξουν όλα αυτά αλλά το κοινοβούλιο θα πρέπει να φροντίσει για αυτού του είδους την ε, υποχρέωση που απορρεύει φροντισει για αυτου του είδου την υποχρεωση που απορρευει συνθηκε για την πρόσβαση στα έγγραφα. Και κάτι άλλο, Πρόεδρε. Κάτι το οποίο δεν το έχω πλήρω καλύψει με την έκθεσή μου. Λέμε ότι στα νομοθετικά έγγραφα θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει για τα διοικητικά έγγραφα να υπάρχει σαν κανόνα στο ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Τα άρθρα που δικαιολογούν την εξαίρεση της ελεύθερης πρόσβασης για τα διοικητικά έγγραφα δεν υπάρχουν πια στις συνθήκες. Άρα αυτές οι διατάξεις δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την εξέλιξη των πραγμάτων. Και δεν θα πρέπει να είναι ο κανόνα το απόρριτο των διοικητικών εγγράφων. Άρα, και εν προκειμένου, ο κανόνα είναι η βασική αρχή τη ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα. Ό,τι θέλετε. Τα θεσμικά όργανα υποχρεούνται να διεκπεριώσουν κάθε αίτηση πρόσβαση στα έγγραφα. Δεν υπάρχουν κατηγορίες εγγράφων που αποκλείονται και εξαιρούνται από την υποχρέωση του να δίνει κανείς πρόσβαση στα έγγραφα. Πολλές φορές τα ε, ε, θεσμικό όργανα το κάνουν κάτι αυτό για ολόκληρες κατηγορίες εγγράφων. Αυτά. Τώρα, εδώ είναι και συνάδελφος ε, η Λάουρα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και ελπίζω ότι θα συμφωνεί με κάποια από αυτά που σας ε, εξέθεσα πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ και και το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την κυρία Χάουταλα. Ήταν πολύ σαφή τα όσα μας εξήγησε για το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Από την άλλη μεριά, βέβαια το θέμα είναι περίπλοκο. Θα σας τα πω και αργότερα. Παντού συμφωνώ 100% ότι δηλαδή θα πρέπει τα θεσμικά όργανα να ασπαστούν τον κανόνα που είναι η ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια και στην ακολουθούμενη διαδικασία και στον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις και τις αποφάσεις. Δηλαδή αυτό θα ήταν η αίσια κατάληξη του θέματος για τους Ευρωπαίους. Τώρα, όσον αφορά τα έγγραφα των τριμερών διαλόγων. Σίγουρα, διάφορα έγγραφα για τα πρακτικά θα πρέπει να διέπονται από ελεύθερη πρόσβαση. Πάντως, όσον αφορά τα έγγραφα, τα ίδια, ε, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι ισχύει. Οι διαπραγματεύσει αυτές από τη φύση τους κάποιες φορές πρέπει να διέπονται από το απόρριτο. Όποιος έχει συμμετάσχει σε τριμερείς διαλόγους γνωρίζει καλά ότι όταν συμμετέχουμε εκεί αλλάζει η τακτική μας, η συμπεριφορά μας, Δεν έχουμε αυτά τα περίφημα έγγραφα με τους πίνακες, με τα διαφορετικές εκδοχές του κειμένου, τι προτείνεται, πού συμφωνούμε κλπ. Δεν είναι επόμενο θέμα το να υπάρχει για ένα ζήτημα μόνο ένα έγγραφο. Γιατί όσο προχωρεί η διαδικασία, πολλές φορές αλλάζουν τα πράγματα και όταν διαπραγματευόμαστε, πολλές φορές ε, επίτηδες πιέζουμε σαν τακτική σε ορισμένα σημεία κλπ. Καμιά φορά αποδίδει αυτή η τακτική, καμιά φορά όχι. Οπότε, εάν τα πάντα δοθούν στη δημοσιότητα, ίσως μας οδηγήσει στο να γελιοποιούμεθα. Από την άλλη μεριά έχουμε και τα λόμπι και την επιρροή τους και έχει δίκιο η κυρία Χάουταλα που είπε ότι κατά τις εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις Κάποιοι, κάποιοι καταφέρνουν να αποκτήσουν πρόσβαση στα έγγραφα. Αλλά εγώ το αντιστρέφω. Γιατί κάποιοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. πρέπει να προβλέπετε τι ισχύει. Και ό,τι ισχύει να ισχύει για όλους. Και για Κοινοβούλιο και για Κομισιόν και για Συμβούλιο. Άρα, θα πρέπει να είναι όσο γίνεται ευρύτερη η πρόσβαση. Αυτό δεν σημαίνει πρόσβαση στο 100%. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε ό,τι ε, επιβάλλεται, ούτως ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να μην έχουν υποψίες οι πολίτες για το τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις αλλά θα πρέπει να είναι σαφές τι δεν επιδέχεται δημοσιοποίηση. Πολλές φορές κάποια έγγραφα μπορούν να δοθούν στη δημοσιότητα όταν κλείσουν διαπραγματεύσεις και πριν από λίγα χρόνια. Συζητήσαμε το τι πρέπει να περιληφθεί σε κάποια έκθεση όταν τελείωσε η διαπραγμάτευση. Θυμάμαι ότι είχαμε ένα σωρό λόμπι που ήρθαν σε επαφή με τον εισηγητή Αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας, δεν γίνεται συχνά, είναι σπάνιο. Οπότε θα πρέπει πρώτα πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι συμφωνήθηκε θα τηρείται. Και ότι θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να αναλύσουμε τι μπορεί να εγκριθεί και τι μπορεί ε, χωρίς πρόβλημα να δημοσιοποιηθεί. Και από την μεριά τι θα πρέπει να παραμείνει σε εμπιστευτικότητα μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσει ε, και όλα να είναι φόρα παρτίδα γιατί αυτό θα καταστρέψει την ουσία της διαπραγμάτευσης. προσευχή πίεση και όπως ξέρετε δεν ωφελεί. Ξέρουμε τι γίνεται με όλα αυτά τα mail που παίρνουμε. Τέλος να τα προχωρήσουμε και ελπίζω τελικά να το βρούμε για να υπάρχει ένα συμβασμός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ε, οι παρουσιάσεις αυτές και η κυρία Χάουταλα θεωρώ πως ανέφερε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, ωστόσο έχω κάποιες ερωτήσεις. Πώς δηλαδή μπορούμε αυτήν την διαφάνεια να την εφαρμόσουμε, να την ε, δημιουργήσουμε έτσι ώστε να έχουμε και την πρόσβαση στα έγγραφα μετά τους ε, τριμερείς διαλόγους. Ε, να σας πω ότι σκέφτομαι. Σκέφτομαι πως αυτή τη στιγμή έχουμε τακτικές ενημερώσεις από τους εισηγητές εδώ στην Επιτροπή σχετικά με την πορεία των τριμερών διαλόγων, όμως τις περισσότερες φορές είμαστε γρήγοροι, ε, τα περνάμε λίγο βιαστικά τα πράγματα και δεν έχουμε αυτή την ακρίβεια που χρειάζεται. Και πολλές φορές συμβαίνει ότι στην ε, Επιτροπή συζητούμε αρκετά, στις ομάδες εργασίας αρκετά. Όταν όμως έρθει η ώρα που μία έκθεση φεύγει από εμά και περνάει στον τριμερή διάλογο, χάνουμε ε, την, ε, τον έλεγχο. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προτείνω κάποια συγκεκριμένη λύση, ε, όμως σίγουρα πιστεύω πως χρειάζεται πολύ περισσότερη διαφάνεια στα έγγραφα, πρόσβαση σε αυτά. Πολλές φορές όμως Αναρωτιέμαι ποιο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ε, πορεία αυτών των εγγράφων όταν φύγουν από εμάς. Ποιο δηλαδή ε, φροντίζει έτσι ώστε να εμείς έχουμε την πρόσβαση σε αυτά, εμείς να ενημερωνόμαστε, διότι μην ξεχνάτε πως εκπροσωπούμε και τους πολίτες που μας ψήφισαν και έχουμε καθήκον απέναντι σε αυτού. Και Υπάρχουν σίγουρα, ε, να, να το γνωρίζετε αυτό, κάποιοι που εποφελούνται από την έλλειψη πληροφόρησης και γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο, ε, στον καλύτερο έλεγχο της ε, πορείας. Δεν μπορώ να σας προτείνω μια γενική λύση που θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε παντού, όμως θέλω να τονίσω αυτήν την ε, διαδικασία που είναι προβληματική και πρέπει, εάν θέλουμε να εφαρμόζεται σωστά ε, η ε, διαδικασία, να βρούμε τα αδύναμα σημεία και να εντοπίσουμε και εκείνους που επωφελούνται από την έλλειψη πληροφόρησης και τις καθυστερήσεις. Ευχαριστώ. Εσείς Φεράρα. Η κυρία Φεράρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξετίμησατε όντω την έκθεση της συναδέλφου Χαουτάλα και συμφωνώ απολύτως με, την, με το περιεχόμενό της, κυρίως όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους, το αρχείο για ενία πρόσβαση για όλα τα θεσμικά όργανα, επίσης ε, την διαφάνεια για τις ομάδες πίεσης στα λόμπι. Όπως αναφέρθηκε εγώ είμαι υπεύθυνη από πλευράς της ΛΥΜΠΕ για την ε, σύνταξη εκθέσεως και υπάρχουν στοιχεία τα οποία αναφέρω και εγώ στη δικιά μου ε, έκθεση. Ας ξεκινήσουμε από τους τριμερούς διαλόγους. Κατά την ε, άποψή μου είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλώς θέμα αρχής, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικαιροποιείται. Και η ταχύτητα και η σκοπιμότητα να προωθούνται αυτές ε, οι πρακτικές, οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να ζημιώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ε, κυρίως τα λόμπι και όχι οι ε, πολίτες ίσως ε, θα διαβάζουν τα έγγραφα αυτά, αλλά η υποχρέωσή μας είναι να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες μας να διαβάζουν τα έγγραφα αυτά. Να σας πω ότι η έκθεση για το προσχέδιο δηλαδή ε, για την πρόσβαση, τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα ε, ανέβηκε στο ίντερνετ έτσι ώστε όποιος ήθελε να μπορεί να τη διαβάσει και να υποβάλει κάποια σχόλια. Εγώ μέσα σε 15 μέρες έλαβα περίπου 150 σχόλια, άλλα καλύτερα, άλλα χειρότερα. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει κινήσαμε κατά κάποιο τρόπο την περιέργεια ε, ε, πολιτών που δεν ε, είναι γνώστες απαραίτητα του θέματος ή δεν είναι συμμετέχοντες στην νομοθετική διαδικασία όπως εμείς, αλλά πάντως το γεγονός ότι θέλησαν να συμμετάσχουν με ικανοποίησε ιδιαίτερα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι από τη στιγμή που μιλάμε για διαφάνεια υποχρεούμεθα όχι μόνο να ε, θεωρητικά να κάνουμε κάτι, αλλά να το κάνουμε και στην πράξη. Όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους, βεβαίως είναι ευαίσθητα ε, ζητήματα και ευαίσθητες συζητήσεις. Το ξέρω γιατί συμμετέχω και τώρα ακόμα σε τριμερείς διαλόγους. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με αυτούς φτάνουν ε, γρήγορα και περισσότερο στους λομπίστες και όχι στους πολίτες. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να γίνονται web streamed οι συνεδριάσεις όπως κάνουμε για εδώ ε, ή και να δημοσιοποιούνται ε, ε, τα πάντα, αλλά θα μπορούσαμε ας πούμε να δημοσιοποιήσουμε τα πρακτικά έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα. Οι τριμερείς διάλογοι βεβαίως είναι ευαίσθητοι, είναι διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά ακριβώς γι' αυτό, ακριβώς γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικές ε, διαδικασίες ε, και λόγω ακριβώς του βάρους που έχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης ε, και στη διαδικασία νομοθέτησης, πιστεύω ότι γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει το περιεχόμενό τους να είναι γνωστό στους πολίτες. Υπενθυμίζω το άρθρο 15, αν δεν σφάλω, της ε, συνθήκης ε, που αναφέρεται ακριβώς στην ε, συμμετοχική δημοκρατία και τη συμμετοχή των, και την εμπλοκή των πολιτών. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων γιατί, και όχι μόνο στο τέλος, γιατί εκεί πλέον πρόκειται για ανακοίνωση, για μια πληροφορία που δίδεται επί θεμάτων τα οποία έχουν αποφασιστεί και κλείσει. ενώ η εμπλοκή του και η πληροφόρησή του θα πρέπει να γίνεται πριν ληφθούν οι αποφάσεις όσον αφορά το μητρό διαφάνειας των ε, μελών των λόμπι. Υπάρχει μια διοργανική συμφωνία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου. Ωστόσο αυτό το αρχείο γίνεται σε, ε, καταρτίζεται σε εθελοντική βάση και επομένως όχι όλες οι ομάδες πίεσης και τουλάχιστον όχι οι πιο σημαντικές ας πούμε ε, έχουν καταγραφεί ε, και οπωσδήποτε λείπει και το Συμβούλιο, δηλαδή λείπουν όλες αυτές οι συνεδριάσεις οι οποίες ε, είναι συναντήσεις του Συμβουλίου με τα λόμπις. Δεν έχετε διερμηνία. Α, Επομένως είναι απαραίτητο, λέω, το Συμβούλιο να προσαρμοστεί ε, σε όλα ε, όσα έχουν συμφωνήσει ήδη το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Όχι μόνο όσον αφορά την εγγραφή ε, στο αρχείο αυτό, στο μητρό αυτό, αλλά και στην κοινοποίηση όλων των συναντήσεων των επιτρόπων, των γραφείων, των υπευθύνων γραφείων υπηρεσιών με το, τους λομπίστες. Το τρίτο. Κοιτάξτε, όλα αυτά γίνονται με κάποια σχετική καταχρηστικότητα και δεν ε, υπάρχει σαφής κανόνας. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι βουλευτές ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ε, έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένες πράξεις και όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα Πρόκειται για πράξεις που μας δίνονται σε μία και μόνη γλώσσα, που όμως είναι δύσκολο ε, να τις ε, κατανοήσουμε, γιατί είναι το περιεχόμενο είναι τεχνικό, δεν έχουμε ε, δυνατότητα να έχουμε λεξικό, δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε κάποιον μαζί μας που να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, δεν μπορούμε καν να πάρουμε σημειώσεις και επομένως είναι ε, δύσκολο ακόμα και για μας και επομένως ανώφελο να διαβάσουμε αυτές τις ε, πράξεις. Ε, και πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξαναδούμε αυτού του είδους την προσβασιμότητα γιατί εμείς από τη στιγμή που πρέπει να νομοθετούμε πρέπει να είμαστε σε θέση να κατανοούμε καλύτερα το περιεχόμενο αυτών των πράξεων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να λάβετε λίγο κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ. Καταρχάς πιστεύω πως το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για πρόσβαση στα έγγραφα παραμερίζεται κάπως με αυτήν την άσκηση της εφαρμογής δηλαδή της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες θεσμικές πτυχές αν αρχίσουμε την συζήτηση για το πόσο προσβάσιμα πρέπει να είναι τα έγγραφα των τριμερών διαλόγων στο κοινό, τότε σίγουρα θα πρέπει να ε, φτάσουμε και στις ε, διοργανικές συμφωνίες. Τα θεσμικά όργανα όμως πρέπει να είναι προορατικά, διότι ήδη υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από νομικής άποψης για την πρόσβαση στα έγγραφα. Και πιστεύω πως πάντα πρέπει να τονίζουμε την αποτελεσματικότητα της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν όμως και κάποιες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δίνουν μεγάλη έμφαση στο θέμα της διαφάνειας και της ε, αποτελεσματικότητας δηλαδή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων απέναντι από τη διαφάνεια. Θα αναφέρω μία από αυτές, μία γνωμοδότηση σχετικά με την ε, πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτή η γνωμοδότηση έδωσε μεγάλο βάρος στο πόσο αναγκαίο είναι να γίνει πιο ανοιχτή η νομοθετική διαδικασία. Αυτό αφορούσε το Συμβούλιο, αλλά μπορούμε να το δούμε και για το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν αρκετοί τριμερείς διάλογοι που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω 1500, ας πούμε 1500 τα τελευταία πέντε χρόνια. Και θεωρώ ότι δεν ε, πληρούμε τις προϋποθέσεις της ε, διαφάνειας, δεν τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Συμπληρώνουμε, ολοκληρώνουμε μάλλον τις ε, διαπραγματεύσεις στην πρώτη ανάγνωση. Και ο κύριος Σβίφκα ανέφερε την ε, ευαισθησία του της ε, πληροφορίας, αλλά να, να σας πω κάτι γι' αυτό. Ας πούμε πως υπάρχει ένας τριμερής διάλογος ε, αναθεώρηση της ενομοθεσίας, του κανονισμού για τη βιολογική γεωργία. Η θέση του Συμβουλίου είναι ότι η βιολογική γεωργία στις πιο κρύες χώρες είναι κάτι το αδύνατον, διότι υπάρχει ζήτηση, ε, υπάρχει σύνδεση με το έδαφος ε, και τα κρύα κλίματα δεν μπορεί να έχει απευθεία σύνδεση του φυτού με το έδαφος, διότι θα παγώσει από το κρύο. Από το κρύο. Είμαι αγρονόμος και το λέω εκ το κράτος μέλος το δικό μου όμως δεν μπορώ εγώ να έχω απαιτήσει να κάνει τα δύνατα δυνατά. Υπάρχει λοιπόν μία αβεβαιότητα και μία νευρικότητα. Όμως εγώ ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο τι συζητιέται στο Συμβούλιο. Πιστεύω πως πρέπει να αντισταθμίσουμε την διαδικασία λήψης αποφάσεων με την ε, ανάγκη για διαφάνεια που προκύπτει και από την ε, νομολογία αλλά και από τις ε, εξελίξεις. Εάν λοιπόν ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ή το δικαστήριο καταλήξουν στο ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, πρέπει να είναι ανοιχτά τα έγγραφα, ελπίζω και εμείς να μπορέσουμε επιτέλους να το συζητήσουμε σε βάθος και να μην κάνουμε λάθη στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με τα σχόλιά σας στο σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 23. Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για την αδιαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εισηγητής είμαι εγώ ίδιος. Και όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συντάσσει αυτή τη στιγμή μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας σχετικά με τη διαφάνεια, την λογοδοσία και την ακαιρεότητα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εμείς παρέχουμε γνωμοδότηση μαζί με άλλες επιτροπές και με τη γνωμοδότηση αυτή θα υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Πιστεύω πως ε, με αυτόν τον τρόπο δίνεται μια καλή συνέχεια στα προηγούμενα δύο σημεία τα οποία συζητήσαμε με την κυρία Χάουταλα. Και οι προτάσεις αυτές ε, κυρίως επικεντρώνονται σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο από κωδικοποιημένους κανόνες, κάτι το οποίο έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, στην Επιτροπή αυτή. Ωστόσο, όπως βλέπετε, τουλάχιστον τα σημεία 5, 6 και 7 περιέχουν και άλλες προτάσεις και άλλες ιδέες οι οποίες καλλιεργούν ένα πνεύμα διαφάνειας. Για παράδειγμα, προτείνω να θεωρήσουμε λυπηρή την απουσία ενός κοινού κώδικα δεοντολογίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Διότι η απουσία αυτή δυσχεραίνει οποιαδήποτε εκτίμηση για την ακαιρεότητα του συγκεκριμένου θεσμικού οργάνου. Παρομοίως και για το σημείο 6. Το σημείο 6 απευθύνεται στους εθνικούς ε, αντιπροσώπους του Συμβουλίου όπου αναφέρεται πως ε, καλό θα ήταν να υπάρχει ένας ε, κώδικας δεοντολογίας ο οποίος θα περιλαμβάνει και κυρώσεις και θα αντιμετωπίζει κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για θέματα ακαιρεότητας ή μη χρηστής συμπεριφορά για περιπτώσεις σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης υπάρχουν κάποιες ε, παρόμοιες ε, προτάσεις που ε, θα, μεταφε... τις δώσουμε στο Συμβούλιο αλλά και για την Επιτροπή των Περιφερειών και για την ΕΟΚΕ. Αυτά τα λίγα έτσι εισαγωγικά λόγια για, την, για το σχέδιο γνωμοδότησης και θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας. Η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ έχω την ίδια άποψη με εσά. Είναι μια συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε πιο πριν με την κυρία Χάουταλα. Γι' αυτό και, γι αυτό και εγώ θα ε, πρότεινα να συνδέσουμε όλα αυτά τα θέματα μεταξύ τους, γιατί αλληλοσυμπληρώνονται. Η, το θέμα της ε, πρόσβασης από τους ε, πολίτες στα έγγραφα πρέπει να συζητηθεί επιτέλους και να βελτιωθεί. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια άλλα σημεία βέβαια, διότι εσείς περιορίζεστε στο διοικητικό αστικό δίκαιο, στη διοικητική πτυχή του θέματος, όμως υπάρχουν κάποια θέματα που πιστεύω πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα. Πιστεύω πως ε, υπάρχει μια κόκκινη ε, γραμμή στις ε, γνωμοδοτήσεις μας. Πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προκύπτουν επειδή το Κοινοβούλιο κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά ε, με, την, ε, με τον ανοιχτό χαρακτήρα ναι. του. Έχουμε web streaming, μας παρακολουθούν ζωντανά. Αυτό δεν συμβαίνει το, στο Συμβούλιο όμως και υπάρχει μία έντονη ανισορροπία, μία έλλειψη διαφάνειας, μία ε, αμφισβήτηση της ακαιρεότητας των θεσμικών οργάνων. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν προβλήματα, κυρίως όμως στο Συμβούλιο. Και εδώ πιστεύω πως πρέπει να αναφερθεί συγκεκριμένα. Να αναφερθεί επίσης και η έλλειψη διαφάνειας των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουμε καμία πρόσβαση σε αυτές τις συνεδριάσεις και στα συνοδευτικά τους έγγραφα και εδώ πιστεύω πως πρέπει να δημιουργηθούν να δημιουργηθεί μια αφετηρία έτσι ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ε, πληροφορία στις συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν. Επίσης, ε, πιστεύω πως πρέπει να αναφερθεί και η εσωτερική ακεραιότητα των θεσμικών οργάνων, διότι είναι έργο μας ως ευρωβουλευτές να ασκούμε ε, τακτικούς ελέγχους και τακτική αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας, ιδιαίτερα για οικονομικά ζητήματα των μελών των θεσμικών οργάνων. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό και δεν είχαμε πολλά δικαιώματα. Κατά την τελευταία νομοθετική περίοδο υπήρχε μια, ε, υπήρχε, υπάρχει, ξέρετε, η δήλωση των οικονομικών συμφερόντων, η οποία δεν έχει συμπληρωθεί από όλους. Εδώ πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων να ε, επικαιροποιηθεί και να βελτιωθεί. Υπάρχουν βέβαια διάφορες κατηγορίες ε, εισοδημάτων των ε, μεσαίων, των υψηλών. Εδώ πιστεύω πως στην περίπτωση εισοδημάτων πάνω από 10.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά, περισσότερα δικαιολογητικά. Από ένα δηλαδή Επίσης, από ένα χρηματικό ποσό και πάνω θα πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις και περιορισμοί ε, στο τι μπορού, μπορεί να κερδίσει κάποιος ε, ασκώντας παράλληλη δραστηριότητα. Η δική μας Επιτροπή ως Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει σημαντικές προσθήκες ιδιαίτερα για όσους καταγγέλουν παρατυπίες, για τους whistleblowers. Ε, μου λείπει μία αναφορά σε αυτούς και πιστεύω ότι η γνωμοδότησή μας πρέπει να αναφέρεται τόσο στους καταγγέλλοντες παρατυπίες όσο και στην προστασία τους. Ευχαριστώ. Κύριος Ράντεφ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα να συγχαρώ τον κύριο Σπόμποτα για την έκθεσή του. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ότι έχουμε σπερμία διατάξεων για τη χρηστή διοίκηση, οπότε και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει το σύστημα να γίνει πιο συνεπές. Χρειάζεται ένας ε, καινούριος κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Αυτό θα διευκόλυνε το πώς θα εφαρμόσουμε τα δυσβασικέ αρχέ, ε, αρχές όπως το δικαίωμα στην χρηστή διοίκηση, αναλογικότητα, κεραιότητα ε, κλπ. Μα πρέπει να υπάρχει μια σωστή δομή για όλε αυτέ τι διοικητικέ διαδικασίε, οπότε θα ήταν πιο αποτελεσματική και η διοίκηση και αντιστοίχω θα ήταν πιο εύκολο να απολαύουν των δικαιωμάτων του ε, οι Ευρωπαίοι πολίτε, το δικαίωμα στην χρηστή διοίκηση και επίση θα μάθουν καλύτερα τα δικαιώματά του και θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε ό,τι οι που προβλέπονται περισσότερο και καλύτερα. Σα ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Κυρία Χάουταλα. Χωρίς μικρόφωνο. Έχει σχέση η δική σας έκθεση με την ε, δική μου, αλλά επίσης και με την επόμενη που θα αφορά ε, τη, διοικητική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η τωρινή σας ε, έκθεση ε, α, έχει αρμοδιότητα η ΑΦΚΟ. Είναι όμως ε, η πιο σφαιρική έκθεση γιατί καλύπτει όλες τις πλευρές της ε, ακαιρεότητα, διαφάνειας, λογοδοσίας στο ύψος υπομένως των προσδοκιών που είπαμε ότι θα καλύψει ευρύτερα την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα και θυμάμαι ότι έχουμε κάνει και κάποιες ακροάσεις στην Επιτροπή μας άρα τέλεια μην Άρα μονεύετε εδώ και την ανάγκη για να υπάρχει ένας κώδικας διοντολογίας και στο Συμβούλιο. Δεν νομίζω το έχουν προσέξει από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον. Και έτσι υπενθυμίσατε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια νοοτροπία που να διέπεται από τέτοιε αρχέ ώστε να επιλύονται και να έρονται οι περιπτώσεις σύγκρουση συμφερόντων. Πολύ καλά τα λέτε. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια. Θα προσπαθήσω ότι μου προτείνετε να το καλύψω παρόλα αυτά. Δεν ξέρω. Όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα, ε, τελευταία φορά τα συζητήσαμε και άλλη φορά στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν πρέπει τώρα να μπουν σε αυτή την έκθεση, γιατί ε, όπως αντιλαμβάνομαι, δεν έχουμε φτάσει ε, σε κάποια συμπεράσματα για το τι θα πράξουμε. Άρα διστάζω σε αυτό το σημείο. Πρέπει να έχουμε κάποιο είδους προσέγγιση ε, συνεπή και να μην πούμε κάτι τώρα από το οποίο θα το άρουμε στη συνέχεια και θα το πάρουν πίσω επομένως θα πρέπει να βρεθεί κάποια διατύπωση ευέλικτη για να καλύψουμε αυτό που είπατε. Ευχαριστώ για όλα όσα είπατε οπότε. Έτσι τώρα κλείσαμε με τα θέματα του πρωινού μας. Το απόγευμα ο κύριος Καβαντά θα προεδρεύσει. Γιατί δυστυχώς έχω κάποια άλλη υποχρέωση. Σας ευχαριστώ πολύ.